Μπορούμε να εστιάσουμε στην ένταση των επιθέσεων παραπληροφόρησης. Επίσης, ε, θα συνεργαστούμε με τον ΝΑΤΟ για αυτό το θέμα. Και θα εξετάσουμε και τις προθέσεις. Πρέπει λοιπόν να είμαστε συντονισμένοι και στοχευμένοι. of the digital ε, θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ποια ε, είναι, πώς θα γίνει η ψηφιακή μετάβαση. Από τη μια πλευρά είναι κάτι το φανταστικό για τον κόσμο, αλλά θα πρέπει να δούμε και τους κινδύνους. Κοιτάξτε, είτε μπορεί να ξεκινεί κανείς ανθρωπιστική βοήθεια, και να βοηθήσεις τους ανθρώπους να ζουν ασφαλώς και υγιώς, αλλά δεν μπορείς να λύσεις γενοκτονία οργανωμένη ανθρωπιστική ε, κρίση. Δείτε τι έγινε με τους Ραχίνγκα. Επίσης ε, βλέπουμε και τις περιπτώσεις όπου ξεκινάνε επαναστάσεις. Μεϊντάν στην Ουκρανία, Φερρυπίν, ξεκίνησε στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι ασπρόμαυρη εικόνα δεν υπάρχει καλό και κακό ξεκαθαρό. Πρέπει να υποστηρίξουμε τα καλά πράγματα, αλλά να αντιμετωπίσουμε και κινδύνου. Τώρα, βάσει των σχολείων σα για τον προπολογισμό, για την υποτίμηση του υπολογισμού, αυξήσαμε τον προπολογισμό τη Stratcom και των διαφόρων μονάδων των αρμοδίων για την καταπολέμηση της ε, παραπληροφόρησης. Πρέπει να βελτιωθούμε όσον αφορά την αναλυτική εργασία, να υποστηρίξουμε την έρευνα, να έχουμε καλύτερο εντοπισμό και καλύτερη εκπαίδευση. Δεν... Έχουμε κάτι πολύτιμο πέρα των χρημάτων. Ξεκινήσαμε συνεργασία μεταξύ θεσμών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κρατών μελών, με τις πλατφόρμες, με τις κοινωνίες των πολιτών και με την έρευνα. Σωστά το είπατε. Χρειαζόμαστε καλύτερη τεχνολογία εντοπισμού και ανάλυσης της παραπληροφόρησης ε, που μπορεί να βλάψει τις κοινωνίες μας. Πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τις ε, εκλογές και να είμαστε σοβαρότατοι ε, μέσω τη σωστή χρήση του GDPR. Έχει προγραμματιστεί για να προστατεύονται τα ιδιωτικά στοιχεία των ψηφοφόρων. Δεν θέλουμε να επαναληφθεί το φαινόμενο Cambridge Analytica. Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Διαφάνεια τη χρηματοδοτήσεω των προεκλογικών εκστρατιών έχουμε υποχρέωση να εγγυηθούμε το ότι στα κράτη-μέλη μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δούμε ε, το φαινόμενο οι τελευταίες εκλογές που έγιναν οι τελευταίες ελεύθερες. Mm. Πρέπει να εγγυηθούμε ότι θα έχουμε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές που θα διεξάγονται. Δεν, θα πρέπει να κερδίζουν σε εκλογές αυτοί που, λένε, που ψεύδονται καλύτερα, αλλά ναι, ούτε αυτούς που χρησιμοποιούν βρώμικες μεθόδους και βρώμικο χρήμα. Ε, αυτό θα πρέπει να το πολεμήσουμε συνεργαζόμενοι. Έχω πολλά άλλα σχόλια, αλλά έχω ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο μου. Ευχαριστώ. Προσβλέπω συνεργασία. Ευχαριστώ την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε και τώρα εκ μέρους του Συμβουλίου ε, η κυρία Τουκάινεν αξιότιμε του Πουράινεν. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση που είναι ένα πραγματικά επίκαιρο θέμα ε, και είναι επίσης και θέμα προτεραιότητας για τη δική μας την Προεδρία. Πράγματι, είναι υποχρέωσή μας να μην υφιστούμε προσπαθειών για να προστατεύσουμε τις εκλογές μας, τη δημοκρατία μας από εξωτερικές παρεμβάσεις με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ελευθερίας του λόγου, ε, των μέσων ενημέρωσης. Ε, αναφερθήκατε πολύ στην επιρροή της Ρωσίας και βεβαίως λαμβάνουμε υπόψη μας την ανησυχία. Υπάρχουν κακόβουλοι ε, φορείς και όπως ε, αυτά που αναφέρθηκαν για τη Ρωσία και οδήγησε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου το Φεβρουάριο αυτού του έτου. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε οριζόντια πέρα από σύνορα, πέρα από φορεί, να μαθαίνει ο ένα από την άλλον με την ανταλλαγή πληροφοριών και με βέλτιστες πρακτικέ. Παρότι λοιπόν έχει σημειωθεί πρόοδος, θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Προσβλέπουμε στην, στο πρόγραμμα δράση Ευρωπαϊκή Δημοκρατία που θα παρουσιάσει η Επιτροπή. Χαιρόμαστε που θα συνεργαστούμε με εσά και με εσά ε, κυρία Γιούροβα για να προχωρήσουν οι πρωτοβουλίες που θα προταθούν. Και πάλι σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση. Και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική ε, σχετικά με τις εξελίξεις στην Ανατολική Γειτονία. Και θα ήθελα να ε, καλωσορίσω θερμά την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Μογκερίνη, και επειδή μάλλον είναι και η τελευταία φορά που ε, έχω εγώ την Προεδρία ενώ εσείς θα έχετε το λόγο και θα είσαστε παρούσα. Ε, δράτω με τις ευκαιρίες για να σας ευχαριστήσω θερμά για όλο αυτό το χρόνο που δαπανίσατε, που περάσατε εδώ κοντά μας, παρότι είχαν και, είχατε και πάρα πολλές άλλες υποχρεώσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη δουλειά σας και για την παρουσία σας στο Κοινοβούλιο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και για τα πολύ ευγενικά σας ε, λόγια. Νομίζω ότι είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που λέω ε, αντίο ε, στην Ολομέλεια είτε εδώ είτε στις Βρυξέλλες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ για την τελευταία φορά που θα είμαι εδώ με το αξίωμά μου, αλλά θα είμαι παρούσα και σήμερα τη νύχτα και αύριο και μεθαύριο, μέχρι την τελευταία στιγμή που θα μπορώ να είμαι εδώ. Θέλω να το εκλάβετε ως ε, ένα ε, μήνυμα αφοσίωσης εκ μέρους μου και αναγνώρισης των προσπαθειών του Κοινοβουλίου στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Με αυτή τη συζήτηση ευχαριστώ πολύ και για την ευκαιρία που μου δίνετε να εξετάσουμε το τι κάναμε τα τελευταία πέντε χρόνια με τους ανατολικούς εταίρους μας. Το 2014, όταν ανέλαβα, τότε ήταν το σημαντικότερο στοιχείο της ε, εξωτερικής πολιτικής μας και της πολιτικής μας ασφαλείας. Και τώρα είμαι περήφανη που μπορώ να σας πω ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθαμε πιο κοντά και στους έξι ανατολικούς μας εταίρους με διάφορους τρόπους και νομίζω μπορέσαμε να βελτιώσουμε ε, την κατάσταση όλων αυτών των κρατών και μέσα από τη συνεργασία. Βεβαίως και παραμένουν κάποιες προκλήσεις, αλλά θα ήθελα σύντομα να παρουσιάσω ε, τα θετικά αλλά και τα αρνητικά στοιχεία, τις αδυναμίες μας, εκεί όπου πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Πιστεύω ότι ο επικοδομητικός αυτός δρόμος που ακολουθήσαμε κατέστη δυνατός γιατί η δουλειά μας εστιαζόταν πάντα στα κοινά συμφέροντα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ανατολικούς εταίρους. Έχουμε τους λαούς της Ευρώπης είτε ζουν μέσα είτε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα 20 ε, θέματα που αφορούν την ανατολική γειτονία. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι, η θέση απασχόλησης, ε, η εκπαίδευση, η ισχυρή κοινωνία των πολιτών, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Θέματα τα οποία βρίσκονται πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη των πολιτών μας. Φέτος είχαμε συμφωνίες εμπορικές με την Γεωργία, τη Μολδαβία, οι πολίτες αυτών των χωρών μπορούν τώρα να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί βίζα όταν έρχονται για δουλειές, για ε, ταξίδι για να επισκεφθούν την οικογένειά τους. Επίσης ε, έχουμε προχωρήσει και στον ψηφιακό τομέα, αλλά πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά στο κράτος δικαίου, στη δικαιοσύνη και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Στις αρχές του έτους εορτάσαμε την 10η επέτειο της Ανατολικής Γειτονίας μαζί με τους εταίρους μας και αποφασίσαμε να δρομολογήσουμε μια διαδικασία διαβουλεύσεων για το μέλλον αυτής της συνεργασίας. Έχουμε συγκεντρώσει πάνω από 200 παρεμβάσεις, όχι μόνο από κυβερνήσεις, κυβερνήσεις και κοινωνίες των πολιτών, αλλά και από ακαδημαϊκούς φορείς, από πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές σας τις ε, παρεμβάσεις. Είμαι χαρούμενη που μπορώ πλέον να αφήσω σε εσά ε, και στον διάδοχό μου αυτό το μεγάλο κεφάλαιο επιτευγμάτων, αλλά και ονείρων, φιλοδοξιών, σταθερά αυτά τα θεμέλια για την επόμενη συνάντηση κορυφή ε, και για το μέλλον της ανατολικής γειτονίας. Κάθε μία από τις έξι χώρες έχει βέβαια διαφορετική διαφορετική κατάσταση, διαφορετικές φιλοδοξίες. Γι' αυτό θα ήθελα πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω αυτές τις φιλοδοξίες. Η Ουκρανία έχει αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις ε, γιατί είχαμε την παραβίαση της κυριαρχίας της από τη Ρωσία. Από το 2014 για την Ουκρανία φτιάξαμε το μεγαλύτερο πακέτο υποστήριξη στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επενδύσαμε περισσότερο στην Ουκρανία από ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου και κανένας άλλος εταίρος δεν έχει επενδύσει στην Ουκρανία τόσο πολύ όσο το πράξαμε εμείς. Αυτό οδήγησε στο να υπάρξουν ε, χειροπιαστά αποτελέσματα. Σήμερα η Ουκρανία είναι πιο ισχυρή και ανθεκτική χώρα από το παρελθόν. Η νέα κυβέρνηση έχει πιο τολμηρή προσέγγιση στις μεταρρυθμίσεις. Οι πολίτες ε, περιμένουν αλλαγές στο κράτος δικαίου, στον αγώνα κατά της διαφθοράς ε, και στην αντιμετώπιση της απάτης. Τους τελευταίους μήνες είχαμε εξελίξεις και στον τομέα της ασφάλειας, ε, κυρίως ε, χάρη της ε, προσέγγισης της Ουκρανίας. Ε, η τετραμερή της Νορμανδίας υπήρξε πολύ σημαντική. Οι δικές μας οι προτεραιότητες ήταν οι ίδιες και με τους εταίρους, ασφάλεια, καλές θέσεις απασχόλησης, ε, θεσμοί που να μπορούν κανείς να τους εμπιστεύεται. Το ίδιο ισχύει και για την δημοκρατία της Μολδαβίας. Στηρίξαμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, βελτίωση του εκλογικού πλαισίου, διασφάλιση ενός ανεξάρτητου συστήματος λογοδοσίας. Η Μολδαβία έχει νέα κυβέρνηση και πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Όπως πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να στηρίξει μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς με κάθε τρόπο ε, και η δική μας υποστήριξη είναι συνάρτηση αυτών των προσπαθειών. Θα εστιάσουμε κυρίως σε μεταρρυθμίσει για την αντιμετώπιση της διαφθοράς των συμφερόντων και είμαι σίγουρη ότι οι κρατικοί θεσμοί μερικές φορές ε, ε, δεν είναι πολιτικοποιημένη. Στην Αρμενία η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για ουσιαστικέ δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται και στη Συμφωνία Σύνδεσης. Η Αρμενία θεωρεί τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το σχέδιο για να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Ε, πράγματι υπήρξαν μεταρρυθμίσεις και μετά την ε, πολιτική επανάσταση της περσινής χρονιάς ε, Είμαστε λοιπόν σίγουροι ότι και αυτή η συνεργασία θα γίνει στο μέλλον πιο στενή. Αζερβαϊτζάν, συνεχίζεται η δουλειά για να ολοκληρώσουμε νέες συμφωνίες. Θέλουμε μια νέα συμφωνία ε, που να συμβαδίζει με τα διεθνή πρότυπα από τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι και την ε, διαφοροποίηση της οικονομίας. Θα συνεχίσουμε για να υπάρχει ε, ειρηνική λύση της διένεξης του Ναγκόρνο Καραμπάχα. Σε ανώτατο επίπεδο θα είναι διαβουλεύσεις και στηρίζει Στηρίζουμε και τις προσπάθειες ε, διαμεσολάβησης ε, της ομάδας Μίνσκ. Έχουμε βέβαια και έναν ειδικό εντεταλμένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ελληνικό εγχείρημα. Η ειρήνη είναι στο DNA μας, στο γεζόν τέτρου μας. Φτάνει στην ουσία του θέματος, του ποιοι είμαστε. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε τα μάλα σε αυτό το θέμα, γιατί δεν έχουν εξαλειφθεί οι συγκρούσεις από την Ήπειρό μας. αντίον η ασφάλεια ε, μαζί ε, με τα ε, διοικητικά προβλήματα αυξήθηκαν τις τελευταίες μήνες. Γεωργία, Οσετία, Γι' αυτό και εμείς αυξάνουμε την παρουσία μας επιτόπου, γιατί η δική μας υποστήριξη στην κυριαρχία και την ταφική ακαιρότητα της Γεωργίας δεν είναι απλά μία δήλωση αρχών. Είναι τα θεμέλια της καθημερινής συγκεκριμένη μας δουλειάς επιτόπου. Η Γεωργία είναι ένας στενός και αξιόπιστος εταίρος στη γειτονιά μας και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ε, δεν φοβόμαστε όταν βλέπουμε να υπάρχουν κίνδυνοι. Σήμερα υπάρχουν κίνδυνοι στη χώρα μπορεί να υπάρξει οπισθοχώρηση σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Και τέλος, όσον αφορά στη Λευκορωσία, οι τελευταίε κοινοβουλευτικέ εκλογέ ήταν μια χαμένη ευκαιρία για να προχωρήσει η χώρα στα διεθνή πρότυπα. Καλέσαμε τι αρχέ να προχωρήσουν σε εκλογικέ μεταρρυθμίσει. Γνωρίζετε όλοι σα ότι έχουμε διαφορέ με τη Λευκορωσία, κυρίω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαι όμω πεπισμένη ότι ο μόνο δρόμο για να προχωρήσουμε είναι να ολοκληρώσουμε τι προτεραιότητές μα. Αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο, όχι μόνο να δουλεύουμε για τα συμφέροντά μα ε, και στι δύο πλευρέ. Ε, πυρηνική ασφάλεια, παραδείγματο χάρη, αλλά για να αντιμετωπιστεί καλύτερα και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι πολύ σημαντικό για μα. Βάζουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο τη δουλειά μα. Αυτό κάναμε τα τελευταία πέντε χρόνια και με του έξι εταίρου μα, παρότι είναι διαφορετικοί μεταξύ του, με διαφορετική προσέγγιση και πάντα εστιάζαμε στον άνθρωπο και όχι στη γεωπολιτική. Και κλείνω λέγοντα, ε, το έχω πει πολλές φορές, όχι μόνο με τους εταίρους μας ε, στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης, αλλά και με άλλους ακόμα πιο πέρα. Έχουμε εξηγήσει ότι η ανατολική ε, σχέση ε, και εταιρική σχέση είναι για τους ανθρώπους, για να, βελτιωθούν, ε, να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής, τα δημοκρατικά πρότυπα, για να υπάρχει μια πιο ειρηνική Ευρώπη που βασίζεται στη συνεργασία. Και κλείνω τις σύντομες αυτές παρατηρήσεις μου ευχαριστώντας εσάς, το Κοινοβούλιο, για την υποστήριξή σας στη δουλειά μας με τους ανατολικούς εταίρους. Γιατί κυρίως στον τομέα αυτό η δουλειά του Κοινοβουλίου ήταν καθοριστική. Εσείς φτιάξατε τις σχέσεις με τα κοινοβούλια αυτών των χωρών, με τις επισκέψεις σας και αυτό ήταν καθοριστικό ε, συνόδευσε τη δουλειά μας, όχι μόνο τη δουλειά των θεσμών, αλλά και των κοινωνιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο λοιπόν τώρα έχει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, κ. Μακάλιστερ. Κύριε Πρόεδρε, ε, αξιότιμοι ε, συνάδελφοι, Ακούσαμε από την είπατε εκπρόσωπο ότι η ανατολική εταιρική σχέση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να επιτύχουμε την αλλαγή των πρώην αυταρχικών σοσιαλιστικών καθεστώτων προς την κατεύθυνση ε, των δημοκρατικών κρατών με οικονομία της αγοράς, ελεύθερη οικονομία της αγοράς. Υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία θα πρέπει ε, να ακολουθούν την πολιτική μας. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθήσει την πολιτική ολοκλήρωση ολοκλήρωση αυτών των εταίρων και αυτό να είναι στρατηγική προτεραιότητα της επόμενης δεκαετίας. Αυτό ισχύει κυρίως για την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία, με τις οποίες ήδη έχουμε σε βάθος σχέσεις και συμφωνίες σύνδεσης. Δεύτερον, αυτή η διαδικασία ολοκλήρωσης απαιτεί από εμάς μια ξεκάθαρη συνεπή στρατηγική ενεργό υποστήριξη και από την άλλη από τους εταίρους μας απαιτεί σοβαρές προσπάθειες γιατί ισχύει μια αρχή που το έχουμε ε, τονίσει επανειλημμένα εδώ στο Κοινοβούλιο, ισχύει η αρχή more for more. Με τα περισσότερα αποκτά κανείς περισσότερα. Δεν υπάρχει όμως ε, καμία αμφιβολία και less for less ε, ισχύει και αυτό επίσης. Όπως το είπε λοιπόν και η κυρία Ήπατη εκπρόσωπος, στα κίνητρα θα πρέπει να περιοριστούμε στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη, στη δημοκρατία και στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Τρίτον, για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το δυναμισμό που υπάρχει σε αυτές τις χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει και να έχει μια διαφοροποιημένη προσέγγιση. Ε, τα που ε, είπε ο κύριος Κουμπίλιος, Άντριος Κουμπίλιος που βρίσκεται εδώ ε, θα μπορούσε να ξεκινήσει παραδείγματο χάν, μια νέα στρατηγική που να αφορά τις σχέσεις με την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση είναι ένα κομμάτι μακροπρόθεσμη στρατηγική έναντι τη ε, Ρωσία, γιατί οι ε, χώρες αυτές ε, που συνδέονται με την Ευρώπη δίνουν ελπίδα στου Ρώσους ότι μπορούν να υπάρξουν αλλαγέ. Το στόχο αυτό εμεί, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τον διεκδικήσουμε μαζί με την σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να κατατεθούν έγκαιρα πριν από ε, το Συμβούλιο την επόμενη χρονιά. Φρεντερίκα, πραγματικά εκ μέρου τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ήσουν ε, ιδιαίτερα αφοσιωμένη κάθε Τετάρτη καθόσουν εκεί στη θέση σου ε, και συζητούσες με όλους τους συναδέλφους. Γι' αυτό λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική δουλειά που έκανες. Εγώ ε, είμαι εκπρόσωπος του ΕΛΚ, εσύ είσαι από τη σχετική πολυομάδα Είχαμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία. Σου εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Φεντερίκα. Ευχαριστούμε, συνάδελφε, την μπλε κάρτα ε, δεν θα την δώσω γιατί έτσι και αλλιώ μετά από λίγο θα λάβετε το λόγο και σας έχουμε βάλει στον κατάλογο των ομιλητών. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Κάτι Πύρη. Ευχαριστώ αγαπητή κυρία Υπατή εκπρόσωπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, γενικά η συζήτηση αφορά την Ανατολική Εταιρική Σχέση. Να σταθώ πιο συγκεκριμένα επί τη Γεωργία και του Αζερβαϊτζάν, επί δύο χωρών. Θα ξεκινήσω με πρόσφατε εξελίξει που, κατά την άποψη, μα προβληματίζουν για την ομάδα στη Γεωργία γίνονται μεγάλε ματαιρίε στην τυφλίδα, διότι η κυβέρνηση τελικά δεν ανταποκρίθηκε στη δέσμευση να αλλάξει τον εκλογικό νόμο το 2020 και να εφαρμοστεί η πλήρη αναλογική. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε στου ψηφοφόρου Γεωργία και περιμένουμε όλα τα κόμματα Γεωργία τελικά να συμμορφωθούν με αυτή την υπόσχεση. Η Γεωργία έκανε πολύ δρόμο όσον αφορά τη δημοκρατία τα τελευταία χρόνια αλλά η παρούσα πολιτική κρίση κινδυνεύει να δημιουργήσει αστάθεια στη χώρα και αυτό είναι κάτι που η Γεωργία δεν μπορεί να το αντέξει. Περιμένουμε από όλα τα πολιτικά κόμματα να ξεκινήσει διάλογος, θέμα πώς να επιληθεί ε, το πρόβλημα του τωρινό. Αζερβαϊτζάν, που είναι μακριά από, σε επίπεδο δημοκρατίας, Όσο αφορά τη δημοκρατία, η δυναστεία Αλίεφ έχει φρικτό ιστορικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το περασμένο μήνα οι αρχέ Βία διάλυσαν ειρηνικέ διαδηλώσει κομμάτων αντιπολίτευση και ντουζίνε από διαδηλωτέ ε, φυλακίστηκαν, ε, ξυλοκοπήθηκαν. Οι ε, παράνομες παρακολουθήσεις διπλωματών της Ευρωπαϊκής Ενώσης σε ιδιωτικές συνομιλίες με μέλη της και την κοινωνία των πολιτών κάνει τη δουλειά πολύ δύσκολη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά. Και Ίσως να υπάρχει ο φόβος ότι το Αζερβαϊτζάν πάει να γίνει Μόσχα. Ήδη συνέβη αυτό προκαιρού πιστεύω και τώρα βλέπουμε δυστυχώς ε, τα αποτελέσματα και την επιβεβαίωση αυτού. Κυρία Ήπατη, εκπρόσωπη, επίση εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, θέλω να σα ευχαριστήσω για την τελευταία πενταετία. Πάντα ήμασταν υπερήφανοι να σα βλέπουμε επικεφαλή τη υπηρεσία μα εξωτερικών σχέσεων, επικεφαλή τη εξωτερική πολιτική. Σα ευχόμεθα ό,τι καλύτερο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you. Συνάδελφε Αυστρεβίτσιος, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωποι, δεν ε, λέμε αντί ακόμα. Ευχαριστώ από την αρχή για τη συνεργασία που είχαμε με, την, ε, με τους φιλελευθέρους και την ομάδα Ρινιού και προσβλέπουμε ε, στο μέλλον σας. Δεν ξέρω ποια θέση θα αναλάβετε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα διασταυρωθούμε πάλι και θα έχουμε καλή αποτελεσματική συνεργασία. Η, Ανατολική, η πρωτοβουλία την Ανατολική γειτονία επέτρεψε εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να, δημιουργήσουμε, να έχουμε ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια περιοχή συνεργασία και ασφαλεία στα εξωτερικά μα σύνορα, τα ανατολικά σύνορα. Για του εταίρου μα είναι μια ευκαιρία να αποκτήσουν την ευημερία και τη σταθερότητα υιοθετώντα ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ και πρότυπα. Μάθαμε πολλά μαθήματα τα τελευταία δέκα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του ενό, ότι η εφαρμογή προγραμμάτων χωρί προσαρμογή των προγραμμάτων στην πραγματικότητα ανάγκες και προσδοκίες των διαφόρων χωρών είναι κάτι που δεν μπορεί να δουλέψει. Για την επόμενη δεκαετία τη ανατολική εταιρική σχέση πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και αντί να εφευρίσκουμε προγράμματα θα πρέπει να καλούμε του εταίρου μα να συμμετάσχουν σε εκείνα που εμεί ήδη εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ανατολικοί μα εταίροι θα πρέπει να έχουν πραγματική δυνατότητα συνεργασία, να γίνουν συνεταίροι μα, να μπορούν να συμπεριληφθούν στι πρωτοβουλίε μα για το κλίμα, την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τη διασυνδεσιμότητα, την ενέργεια και την κοινωνική ε, συμπερίληψη και κάλυψη των πάντων για τα σχετικά προγράμματα. Είναι προφανέ ότι εκείνοι που καταβάλουν μεγαλύτερε προσπάθειε και παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τι μεταρρυθμίσει που εφαρμόζουν, θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να εμβαθύνουν τι ε, σχέσει του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αρκετές χώρες που χωρίς ε, το, να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσης συμμετέχουν στην ενιαία αγορά. Οι εργάτες της Ουκρανίας ε, συμβάλλουν ε, σε στις οικονομίες της Λιθουανίας, της Πολωνίας και άλλων χωρών και τους αξίζει να προστατεύονται τα εργατικά τους δικαιώματα. Συνάδελφοι, πρέπει να τονίσουμε εκ νέου ότι δημοκρατικά κριτήρια, κυρίως η προσκόλληση στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κάτω δικαίου πρέπει να είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Κύριε Πρόεδρε, Δευτερολογώντα αυτό την ανησυχία τη Κάτι Σπύρι και εγώ εκφράζω ανησυχία για την κατάσταση στη Γεωργία και πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι πρέπει να αντιδράσουμε όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στην Τυφλίδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Και τώρα για δύο λεπτά και δυόμιση λεπτά, Φων Κράμον Ταουμπάντελ. Έχετε το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βλέποντας την ανατολική μας γειτονιά, πολλοί τη βλέ... βλέπουν μια εικόνα σπρώμαυρη. Αυτή η δράση υποστηρίζει τα συμφέροντα της Ρωσίας στην περιοχή ή τους εκπροσώπους της δύση. Αλλά είναι λάθος ερωτήματα αυτά. Οι ηγέτες αυτών των χωρών δεν πρέπει να πιστεύουν σε εμά, πρέπει να πιστέψουν στο μέλλον των χωρών τους. Η Μολδαβία, η Γεωργία, η Ουκρανία, Όλε είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και στις τι περιπτώσεις είδαμε φιλόδοξε κινήσει για μεταρρυθμίσει, αλλά για διαφορετικούς λόγους όμω, σήμερα δεν είμαστε σίγουροι κατά πόσο αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν ή θα καταλήξουν σε μια δημοκρατική διολίστηση. Και το θέμα δεν είναι κατά πόσο οι πολιτικοί μπορεί να γράφουν ωραία ανακοινοθέντα τύπου περί αξιών της Δύσης, όλοι μπορούν, είμαι σίγουροι, Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούν να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις με την που υποστηρίζονται από την κοινωνία τους. Ε, οι... αν οι χώρες της Ανατολικής Γειτονίας περιμένουν να, μας, να τους υποστηρίξουμε, κυρίως εφόσον άλλοι γείτονες εργάζονται κατά ε, των επιτυχιών αυτών των χωρών. Η οικονομική επιτυχία αυτών των χωρών της γειτονίας θα ήταν η μεγαλύτερη ήττα του Πούτιν οι κοινωνίες της Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Μολδαβίας θέλουν να βοηθήσουμε τη διαδικασία μεταμόρφωσης των κοινωνιών αυτών, κάτι που δεν γίνεται χωρίς θυσίες. Ε, γνωρίζω τι θέλω να δω σε αυτές τις χώρες. Ε, δεν, υπερασ... δεν προωθώ ε, τις μεταρρυθμίσεις διότι θα εξυπηρετήσουν γεωπολιτικά συμφέροντα όπως είπατε κυρία Μογκερίνη ή την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Θέλω να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις διότι η συντριπτική πλειοψηφία των λαών που ζουν εκεί θέλουν να δουν δημοκρατικές και ευημερούσε κοινωνίες. Μια οικονομία που εργάζεται για τον κόσμο και όχι για τους λίγους ολιγάρχες. Ένα κράτος που υπηρετεί τους πολίτες και όχι τους πολιτικούς και τα συμφέροντα των πολιτικών. Για μια αλλαγή που έχει νόημα χρειαζόμαστε ισχυρέ κυβερνήσει αφοσιωμένε αυτό το σκοπό. Όμω, μια ισχυρή κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει εκτελεστική εξουσία ανεφελέγχου. Είναι ανησυχητικό που βλέπουμε αυτές τις τάσεις στη Γεωργία και στην Ουκρανία, κάτι που ήδη αναφέρθηκε. Όμως οι κυβερνήσεις δέχονται πίεση, αλλά που δεν πρέπει να απειλούν ή να καταπιέζουν την κριτική. Ε, Εμεί δεν επικρίνουμε κάποιον αν είναι υπέρ Βρυξελών, υπέρ του Κρεμλίνου. Εμεί θέλουμε να είναι, δημο... αν είναι, βλέπουμε αν είναι κάποιο δημοκρατικό και αν υποστηρίζει δημοκρατικού θεσμού ή όχι. Και ναι, θέλει ο Πούτιν να έχει πολιτικού που μπορεί να εξαγοράσει και να επηρεάζει ο Πούτιν. Εμεί δεν έχουμε αυτό το στυλ. Θέλουμε να θέλουν ηγέτε μεταρρυθμίσει, θέλουμε να έχουμε ε, θεσμού που λειτουργούν, αυτό είναι προ μα, να λειτουργούν χωρί ε, τον Πούτιν, χωρί του ολιγάρχε και χωρίς εμάς ακόμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπαθεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα της διεύρυνσης προς Ανατολάς. Ας δούμε λιγάκι τι γίνεται στην Ουκρανία. Η Ουκρανία εδώ και χρόνια έχει ε, τραβήξει πάνω της ε, τη μεγαλύτερη προσοχή, κυρίως λόγω της αντιπαράθεσης της με τη Ρωσία. Από το 2014 στην Ουκρανία επενδύθηκαν 14 δισεκατομμύρια ευρώ με τη μορφή δανείων και επιχορηγήσεων για να στηριχτούν οι μεταρρυθμίσεις. Και μεταξύ αυτών και η δικαστική μεταρρύθμιση για να πλησιάσει αυτή τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και εκεί εντάσσεται και η εφαρμογή της Συμφωνίας ΧΚΙ σχετικά με την απαγωγή παιδιών. Εάν ε, απάγεται ένα παιδί ε, σε μια χώρα που έχει υπογράψει αυτή τη συμφωνία, συγκεκριμένα τώρα στην Ουκρανία, τότε οι δικαστικές αρχές οφείλουν να μεριμνήσουν έτσι ώστε το παιδί να επιστρέψει ε, εκεί από όπου απήχθη. Η Ουκρανία όμως δεν τα εφαρμόζει όλα αυτά. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες ειδήσει για ευνοιοκρατία, ε, για διαφθορά. Μέχρι τώρα υπήρξαν 33 ε, περίπου απαγωγές παιδιών. Ο τότε Υπουργό Δικαιοσύνη ομολόγησε σε μία συνέντευξη ότι κανένα από τα παιδιά δεν επιστράφηκε στη Γερμανία, αν και αποφάνθηκαν διαφορετικά τα δικαστήρια τη Ουκρανία. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ καλώ την Ουκρανία αυτή τη συμφωνία τη Χάγη επιτέλου να την εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν το κάνει αυτό η Ουκρανία, δεν θα τη δώσει πια δάνεια και επιδοτήσει μέχρι να γυρίσουν επιτέλου τα παιδιά εκεί που πρέπει να επιστρέψουν κυρία παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία, είπατε εκπρόσωπη, σας ε, ευχαριστώ για τα τελευταία πέντε χρόνια συνεργασίας και καλή σας ε, επιτυχία. Η υποστήριξή μου για τα έθνη της, της ανατολικής εταιρικής σχέσης είναι αμετάκριτη εφόσον ε, δούλεψα και στο το τμήμα εξωτερικών της δύο θέματα είναι σταθερά εκεί. Το ένα είναι ο σταθερός δυτικός προσανατολισμός των κοινωνιών και η βούλησή τους να μείνουν εδώ μαζί μας και ο δεύτερος είναι, σταθερός παράγοντας, είναι η βούληση της Ρωσίας να τους υποτάξει και να τους αποσταθεροποιήσει παρά τις προσπάθειές μας ε, εξακολουθούν να ε, υφίστανται δύσκολα ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Πολλά ε, δυναμικά και θετικά στοιχεία έχουμε. Έχουμε επιτυχίες στις πολιτικές μας βέβαια, αλλά υπάρχουν και κάποια ζητήματα που μας προβληματίζουν. Η Ουκρανία είναι ακόμα υποκατοχή τα λιμάνια της θάλασσας Αζόφ ακόμα είναι μπλοκαρισμένα. Υπάρχουν ε, ε, κρατούμενοι στις ρωσικές φυλακές. Στην Γεωργία είναι μια πραγματική ανησυχία που ανησυχούμε πάρα πολύ για τις τελευταίες εξελίξεις. Πιστεύω πως η πολιτική κρίση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και πρέπει να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε οι ε, σχέσεις της ε, ανατολικής γειτονίας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις. Ε, κλιματική αλλαγή, φτώχεια στην ενέργεια, δεν μπορούν να χειριστούν μόνοι τους τους πόρους τους, δεν μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, να ξεπεράσουν επίσης και το παρελθόν. Αυτά ενδεικτικά τα αναφέρω. Αλλά και το θέμα του εκδημοκρατισμού της κοινωνίας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική μας προς τις χώρες αυτές αποκινούμε τους πολίτες των κρατών πρέπει να συνεχιστεί και αυτό σημαίνει περισσότερο κράτος δικαίου, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, συμπερίληψη της κοινωνίας των πολιτών, να μπορούν ε, οι παράγοντες να παρεμβαίνουν στις κοινωνικές εξελίξεις, προσπάθειες για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, δημιουργία δημοκρατικών θεσμών, προαγωγή του δημοκρατικού διαλόγου, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη, διαφάνεια, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, ειρηνική διευθέτηση ε, αντιπαραθέσεων και ε, πιο συγκεκριμένα έχουμε το παράδειγμα της ε, Μολδαβίας. Η εκλογή ε, του τελευταίου πρωθυπουργού ήταν μια κάποια αχτίδα φωτός όταν προτάθηκαν οι υποψήφοι για τη θέση του εισαγγελέα οι ε, σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ε, κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας ε, που δυστυχώς κατέληξε σε παρέτηση της κυβέρνησης. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι η Μολδαβία έχει επιστρέψει σε σκοτεινές πρακτικές που χαρακτήριζαν την προηγούμενη κυβέρνηση. Ο Βλαντιμίρ Πιανούκ, ο ολιγάρχης, είναι στην εξουσία και η Ωνά Ροζάτσι και ο Πετρέγκο, οι ακτιβιστές, διώκονται ποινικά. Εγώ λοιπόν ε, επιθυμώ από κοινού να σκεφτούμε το πώς ακριβώς ε, θα μπορέσουμε στις ε, χώρες μας να στηρίξουμε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε αγαπητές συνάδελφε. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κουμπίλιους Άντριους. Κύριε Πρόεδρε, Κυρία ε, είπατε πρόσωπη θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Όλοι κατανοούμε γιατί αγωνίζονται για τη δυνατότητα ένταξη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ουκρανία, η Γεωργία και η Μολδοβία. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε περισσότερο εμείς ε, ε, υπέρ της ένταξή τους από ότι ηγέτες των χωρών αυτών. Σήμερα θα μιλήσω για τη Γεωργία και όχι για τη Μολδαβία που ο Πρωθυπουργό της, ο καινούριο αποφάσισε πρώτη επίσκεψη να πάει στη Μόσχα. Οι πρόσφατε εξελίξει μα ανησυχούν πολύ όσον αφορά το μέλλον τη δημοκρατία στην ε, χώρα αυτή. Καμιά δημοκρατία, καμιά ένταξη, καμιά ολοκλήρωση. Ξέρουμε ότι ε, ο αρχηγό του Σοσιαλιστικού Κόμματο δεν εφαρμόζει την πρόσχεσή του για την ένταξη, την, ε, την του συστήματος ε, της αναλογικής στο εκλογικό σύστημα. Τώρα η εμπιστοσύνη των Γεωργιανών στο Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία έχει χαθεί δεν ε, τήρησαν την, την υπόσχεσή τους, ίσως γιατί φοβούνται να μην χάσουν τις εκλογές ε, την, ε, την επόμενη φορά. Τι, μπορούμε να... να... τι δίδαγμα μπορούμε να αποκομίσουμε. Ίσως ότι το κυβερνών κόμμα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα παλιά κόλπα για να ξανακερδίσει τις εκλογές. Αυτή η συζήτηση είναι καλή ευκαιρία για να παροτρύνουμε τους ηγέτες της Γεωργίας να μπουν σε πραγματικό και καρποφόρο διάλογο με την αντιπολίτευση. Επίσης θα πρέπει το κυβερνών κόμμα μαζί με την αντιπολίτευση να συμφωνήσουν στη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος γιατί ο κόσμος δεν το εμπιστεύεται αυτό το σύστημα. Το γερμανικό σύστημα θα μπορούσε να αποτελεί τη βάση για μια τέτοια συμφωνία γιατί δεν απαιτεί κιόλα αλλαγή του Γεωργιανού Συντάγματο. Τέλο, το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να παροτρύνει τα νόμιμα κόμματα να εφαρμόσουν ε, νέο εκλογικό σύστημα και να πάψει η πρακτική της επιρροής της εκλογές. Να βοηθήσουμε τη Γεωργία με αυστηρή κριτική. Μάλιστα, ευχαριστώ. Τώρα το λόγο ο κύριος Πίτσουλα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τα πέντε χρόνια αγαστής συνεργασίας και να σας ευχηθώ ε, ό,τι καλύτερο ε, για το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε στενότερους δεσμού με τις γειτονικέ χώρες όπου έχει συμφέροντα για την ενέργεια και για ολοκληρωμένες εμπορικές σχέσεις, αλλά και για να αυξήσει την επιρροή της. Εμείς παρατηρούμε τις εξελίξεις αυτές τι χώρες ε, που επηρεάζουν όμως αυτά τα ε, σχέδια, ενώ ε, σχεδιάζεται μια διάσκεψη κορυφής στην Νορμανδία. Δυστυχώς στη Γεωργία υπάρχει ένα νέο κύμα αστάθειας. Στην Λευκορωσία οι εκλογές διαρκώς ε, αποτυγχάνουν συντήρηση διεθνών προδιαγραφών. Στη Μολδαβία ο κυβερνητικός συνασπισμός διαλύθηκε. Στην Αρμενία τα πράγματα φαίνονται σταθερά, εκτός από τη μόνιμη σύγκρουση με το Αζερβαϊτζάν. Θέλω δεν αναφέρω και τις σχέσεις της Ένωσης με το Αζερβαϊτζάν όπου η ηγεσία είναι, μιλά ξεκάθαρα ενάντια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γεωπολιτικές προκλήσεις και περιστάσεις σε αυτές τις χώρες απαιτούν ισχυρότερες και στενορότερες ενέργειες από πλευράς Ένωσης. Η επερχόμενη διάσκεψη κορυφής θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν να ενισχύσουμε τις γεωπολιτικές μας φιλοδοξίες. Ο κύριος Πάετ τώρα. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω τη Φεντερίκα Μογκερίνη, άριστη συνεργασία μας. Η ανατολική εταιρική σχέση πρέπει να παραμένει ψηλά στην ατζέντα του Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Πρέπει να έχουμε σταθερή και ασφαλή γειτονία. Είναι προ όφελο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Πρέπει να εξακολουθούμε να θαρρύνουμε τι χώρε τη Ανατολική Γειτονία να κάνουν τι αναγκαίε μεταρρυθμίσει και να τι βοηθήσουμε. Όμως αυτό που βοηθάει περισσότερο την πρόοδο σε αυτές τις χώρες είναι η επιθυμία της Ρωσίας να τις διατηρήσει στην ε, επιρροή της. Αυτό τις καθυστερεί. Πέντε από τις έξι χώρες εταιρικής σχέσεως έχουν στην επικράτειά τους συγκρούσεις. Αυτό εμποδίζει τις χώρες από το να προχωρήσουν. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει σαν μία από τις προτεραιότητες την προσπάθεια εξέβρεσης λύσεων σε αυτούς τους παγωμένους ή τόσο, τόσο παγωμένους, ε, τις τόσο παγωμένες συγκρούσεις για να μπορέσουν να αφοσιωθούν αυτές οι χώρες μετά στην ανάπτυξή τους και τις μεταρρυθμίσεις. Είναι επιτακτική ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπιστεί την εδαφική ακαιρεότητα των χωρών τη Ανατολική Γειτονία. Επίση, πρέπει να εγγυηθούμε επαρκή χρηματοδότηση στο νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο για να τι βοηθήσουμε να συνεχίσουμε τα ρυθμίσει. Τακτικό διάλογο υψηλού επίπεδου είναι κάτι αναγκαίο και συγκεκριμένοι στόχοι απαιτούνται για την περίοδο μετά το 2020. Τέλο, ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στη Γεωργία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία που έδειξαν ε, διακαεί πόθο να πλησιάσουν ε, την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πειθαρχία σας όσον αφορά το χρόνο αγόρευσης. Η κυρία Χάουντι Χάουτελ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εμένα είναι χαρά μου να ευχαριστήσω την ύπατη εκπρόσωπο που ήταν τόσο δραστήρια στη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σημείωσα την αυξανόμενη εκτίμησή σας όσον αφορά την κοινοβουλευτική συνεργασία στην εταιρική, την, ε, στη σχέση με τις ανατολικές χώρες, τις ε, χώρες της γειτονίας. Είναι πρόθυμες να συνεργαστούν οι χώρες και η συνεργασία έχει φτάσει σε μεγαλύτερο βάθος όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικής και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με τι χώρε Ανατολική Γειτονία. Είπατε ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα για το κράτος δικαίου και για το δικαστικό κλάδο. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σας, διότι δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε σχετικά με τα τεκτενόμενα εκεί και πιστεύω ότι αυτό που ανέφεραν ήδη οι συνάδελφοι όσον αφορά τι πρόσφατε εξελίξει στη Μολδαβία και τη Γεωργία οφείλονται πολύ στην έλλειψη σταθερότητας των θεσμών Προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε τη δημιουργία θεσμών, αλλά βλέπουμε, Φερρυπίν, ότι στη Μολδαβία η ομάδα του παλιού καθεστώτος, ή μάλλον το, το παλιό καθεστώς έχει αρπαχθει στην εξουσία και κρατειται πολύ καλά και προσπαθεί να προστατεύσει η παλιά εξουσία τα συμφέροντά της. Εάν κάνουμε περισσότερα σε αυτούς τους τομείς στις γειτονικές μας χώρες, νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο να μην φυστούμε προσπαθειών στο κράτος δικαίου και το δικαστικό κλάδο. Είναι ενδιαφέρον το ότι είχαμε μια αιτήσια έκθεση για τη δημοκρατία από την International Idea, ότι στην Ήπειρό μας η μόνη χώρα που έχει βελτιώσει τα δημοκρατικά της πρότυπα τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο χρόνο μάλλον, είναι η Αρμενία και με τα χαράς μεγάλης λέγω ότι οι εξελίξεις στην Αρμενία είναι ένα, φωτιν... είναι ένα φως στην περιοχή Φάρος στην περιοχή πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και υποστήριξη της αντοχής των γειτονικών μας χωρών κατά της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας. Κυρία Χάουταλα, ο κύριος Τζίμνιοκ έχει μια γαλάζια κάρτα. Έχει ερώτηση. Δέχεστε, κύριο Τζιμνιουκ. Μία ερώτηση προς τους δύο προλαλήσανες, αλλά ο ένας έχει φύγει νομίζω. Αυτό το εγχείρημα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ε, αμυγός ε, ελιτίστικο πρόγραμμα και οι πολίτες δεν το θέλουν αυτό, δεν το στηρίζουν. Μόνο στη Γερμανία, με βάση πρόσφατες σφιουμετρήσεις, πάνω από 46% είπαν ότι δεν θέλουν ε, τη διεύρυνση. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό το αγνοείται, γιατί από ό,τι φαίνεται θεωρείται ότι ο λαός είναι χαζός. Θεωρείται ότι, είμαστε, ότι εμείς είμαστε πιο έξυπνοι. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, δεν μιλάμε για διεύρυνση απόψε. Μιλάμε για τη δημιουργία πιο σταθερής και δημοκρατικής γειτονιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος αυτού, όπως εξήγησε και η Πατή Εκπρόσωπος, είναι να αφεληθούν οι λαοί. Και σαν συγκεκριμένο αποτέλεσμα της ε, διαδικασίας είναι η επαλλαγή αποθεώρηση για τους κατοίκους Γεωργίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας δεν είναι ένα ελιτίστικο πρόγραμμα. Ευχαριστώ κύριε Χάτολα. Συνάδελφε, ε, γνωρίζετε πολύ καλά ναι, ότι ναι, ναι. για να υπάρξει κάποιο βήμα διεύρυνσης ε, πρέπει να υπάρχει ομοφωνία και οποιαδήποτε μορφή διεύρυνσης ε, προκύπτει μετά από μια σαφή διαδικασία και συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να γίνονται. Ως εκ τούτου κανείς δεν μπορεί αυθαίρετα να κάνει κάτι, αλλά οι κανόνες θα πρέπει να τηρούνται και από τις δύο πλευρές. Μην ρίχνετε στάχτη στα μάτια μάτια των πολιτών. Το λόγο έχει ζητήσει η κυρία... ο κύριος Μαριάννη Τιερή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κάποια, κάθε χώρα ε, σημειώνεται από την ιστορία της και τα σύνορά της. Και αυτές οι χώρες είναι ταυτόχρονα πρώην σοσιαλιστικές σοβιετικές χώρες που γύρισαν την πλάτη στον κομμουνισμό και χώρες με την εξαίρεση της Μολδαβίας που όλες έχουν ένα σύνορο κοινό με τη Ρωσία. Η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτές τις πραγματικότητες και να μην απαιτεί συστηματικά από τις χώρες αυτές να στρέψουν πλήρως την πλάτη τους προς το παρελθόν τους και την ιστορία τους ε, την τριακονταετή Ευρώπη και, Ευρώπη Ρωσία. Θα θα πρέπει λοιπόν ε, να έχουμε δυνατότητα να φροντίσουμε αυτές οι χώρες να εξυπηρετούν τις συζητήσει ε, μεταξύ των Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ενώσης, να γίνουν γέφυρες. Να ζητάμε να επιλέξουν μεταξύ του αλουνού και του αλουνού, τους οδηγούμε στην καταστροφή. Λυσμονήσαμε λίγο γρήγορα ότι μετά από μια συμφωνία σύνδεση που ζητήσαμε από την Ουκρανία να γυρίσει την πλάτη στην ιστορία, που ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα γεγονότα τα γνωστά ξέσπασαν και οδήγησαν τη χώρα στο χάο. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να μα παρακινεί σε αυτή την περιοχή να είμαστε κάπω σεμνοί και ταπεινοί και να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε στο ρυθμό που ακολουθούν κανονικά αυτέ οι χώρε. Ευχαριστώ κύριε Τζαμπάφσκι, παρακαλώ. Σας, ευ... Σας ευχαριστώ. Είπατε εκπρόσωπε συγχαρητήρια. Ε, θα προχωρήσω για το θέμα του, της ε, ανατολικής ε, εταιρικής σχέσης. Είναι δύσκολο για πολλούς από εμά, αλλά για να, γίνει, για να είναι επιτυχή, θα, επιτυχής, θα πρέπει να έχει στόχο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όταν συζητάμε χώρες όπως το Αζερβαϊτζάν και η Γεωργία, υπάρχουν project που θα πρέπει να εφαρμοστούν με τη βοήθεια της Ένωσης όπως τα project υποδομών, ε, η δημιουργία υποδομών, η κατασκευή υποδομών, ώστε να μπορέσουν οι χώρες αυτές να είναι πιο προσιτές σε μας. Και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, δεν θα μείνουμε σε λόγια. Κατά την προηγούμενη θητεία ακούσαμε πολλά λόγια, όμως τα λόγια δεν ε, βοηθούν. Πρέπει να εστιάσουμε σε πραγματικά απτά αποτελέσματα. Δύο λεπτά τώρα ο Σικώρσκι. Σικόρσκι. Και, πρόεδρε, το 2008 όταν η Πολωνία και η Σουηδία πρότειναν ένα πρόγραμμα ανατολικής εταιρικής σχέσης εμπνευστήκαμε από δύο διαδικασίες. Την Ένωση για την Μεσόγειο, δηλαδή ένα ε, project για την ε, σταθεροποίηση της γειτονίας μας και για το project προετοιμασίας των, χωρών, των πιθανών υποψηφίων χωρών. Δεν ήταν ένα project κατά της Ρωσίας. Η ίδια η Ρωσία αποφάσισε ότι κινδυνεύει από τη δημοκρατία και το ελεύθερο ε, εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε την Ρωσία και ε, και να, ως παρατηρητές τι κάναμε, έχουμε δαπανίσει πάνω από 10 δίσεις σε πολύτιμα ε, project, υποδομές, έχουμε εταιρικέ σχέσεις ελευθέρων συναλλαγών με τις χώρες αυτές. 80.000 νέοι υποφελήθηκαν από το πρόγραμμα Erasmus Plus ε, και όλα αυτά ωστόσο δεν μας βοήθησαν να ιτήσουμε τις μη ανταγωνιστικές δομές των οικονομιών των χωρών αυτών. Καταφέρουμε να φτιάξουμε κάτι σαν την Ένωση για τη Μεσόγειο, αλλά όχι, ε, δεν είναι όλα τέλεια. Ελπίζω ότι η Κομισιόν που εγκρίναμε σήμερα θα δώσει συνέχεια στην Ανατολική Εταιρική Σχέση. Είναι ένα πολύτιμο project που φέρνει πιο κοντά τους ανατολικούς μας γείτονες στα στάνταρ μας. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Καλιουράνα, Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητή Φρεντερίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που έκανες, περισσότερα για, για τη Γεωργία. Όπως αναφέρανε και οι συνάδελφοι, το Γεωργιανό Κοινοβούλιο καταψήφισε τροπολογίες για την εγκαθίδρυση ε, του αναλογικού συστήματος για τις εκλογές του 2020. Ήταν ε, μη αναμενόμενο. Ε, αυτό προκαλεί αναταραχές στην κοινωνία και έφερε τον κόσμο στους δρόμους. Έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους. Θα ήθελα να καλέσω όλα τα πολιτικά ε, κόμματα της Γεωργίας να συγκεντρωθούν να βρουν λύση, ώστε να μην, τεθεί σε κίνδυνο, η να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ελπίδες οι δημοκρατικές του λαού της Γεωργίας. Ακούσαμε τον ε, εκλεγμένη πρόεδρο της Επιτροπής σήμερα που δεν ανέφερε την ε, ανατολική εταιρική σχέση. Αυτό ήταν απογοητευτικό και ως υπεύθυνη για τις σχέσεις με τις χώρες του Νότιου Κάφκασου θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους μου τους ανατολικούς εταίρους για την πλήρη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις ρυθμίσεις και ευρωπαϊκές προσδοκίες αυτών των χωρών. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Κουτσούκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Μογκερίνη. Ε, δράτω με τις ευκαιρίες για να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την ενεργό συμμετοχή σας στο Κοινοβούλιο και σας εύχομαι καλή τύχη για το μέλλον. Η Ανατολική Εταιρική Σχέση έχει στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Μα ενδιαφέρουν πολύ οι εξωτερικές σχέσεις. Σήμερα όμω πρέπει να επανεξετάσουμε την προσέγγισή μα και να βρούμε νέε προτεραιότητε. Έχουν λάβει χώρα σημαντικέ αλλαγέ στου ανατολικού εταίρους. Τα τελευταία χρόνια παρά το παρελθόν Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία έδειξαν ότι επιθυμούν να ε, ενωθούν περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς ε, οι διαδικασίες είναι δύσκολες, ε, η δημοκρατία του είναι εύθρευστη και βλέπουμε και πάρα πολλές διαδηλώσεις στις χώρες αυτές. Βασικό αίτιο είναι ότι υπάρχουν παγωμένες συγκρούσεις στα εδάφη τους. Γι' αυτό λοιπόν καλό τη νέα Επιτροπή να εμβαθύνει σε αυτές τις σχέσεις για να έχουμε ευρωπαϊκές δημοκρατίες σε αυτή την ανατολική γειτονιά μας. Ευχαριστούμε ο κύριος Βατσικόφσκι Γιάννη. Ε, πρόεδρε, αγαπητή Φεντερίκα, μεγάλη μας χαρά να δουλέψουμε μαζί σας ε, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, και εδώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο διάστημα που είμαι Ευρωβουλευτής 30 χρόνια μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού το εγχείρημα της Ευρώπης ε, της ελεύθερης και δημοκρατικής Ευρώπης δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν ακόμα χώρες και υποψήφιες χώρες που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Δέκα χρόνια μετά την ανατολική εταιρική σχέση έχει φτάσει η στιγμή να επανεξετάσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Ε, χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική για την ανατολική εταιρική σχέση. Η νέα στρατηγική της ανατολικής εταιρικής σχέσης ε, υποτίθεται βασίζεται σε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση που θα οδηγήσει στη διεύρυνση ε, δεν πρέπει να φοβόμαστε τη λέξη διεύρυνση. Η διεύρυνση είναι ακρογωνίως λίθος της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και ε, η μακρινή προοπτική της ένταξης αρκεί για να επικρατήσει ειρήνη στη γειτονιά μας. Ε, το να είναι κανείς μέλος, αυτό είναι καταλήτης. Αντίθετα λοιπόν με τον κύριο Μακρόν, εγώ πιστεύω πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή την Ευρώπη και να δεχτούμε νέα μέλη σε αντίθεση με τους υπουλήπους, ο κύριος Μούρεσαν έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Μογκερίνη, ήθελα να μιλήσω για τη δημοκρατία της Μολδαβίας, ένα κράτος στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια φορά μιλήσαμε για τη Μολδαβία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση φιλοευρωπαϊκή τότε έχει αναλάβει τα καθήκοντά της όταν ξεκίνησε την κουβέντα. Ανετράπη η κυβέρνηση μέρου από τα κόμματα τα φιλορωσικά και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί στη Μολδαβία. Είναι κάτι σοβαρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το λέω αυτό διότι αν έχουμε στις πόρτες μας χώρες με κυβερνήσεις φιλοευρωπαϊκής που προσπαθούν να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο ε, υπ' αυτού του όρου θα αυξηθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση στη Μολδαβία ε, επιδεινώνεται Κυρία είπατε εκπρόσωπε, πρέπει να δράσουμε. Υποστηρίζουμε τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις, αλλά δεν αρκούν τα λόγια. Τι θα πρέπει να κάνουμε, καταρχάς να πούμε στους φιλορώσους ποιες είναι οι συνθήκες, οι όροι που θέλουμε. Ο Πρωθυπουργός ο Μολδαβίας πήγε αμέσως στη Μόσχα και πήρε ε, κάποια οικονομική βοήθεια χωρίς διαφάνεια. Αυτή είναι η κανόνες του παιχνιδιού. Αυτοί οι κανόνες του παιχνιδιού θα ε, γίνουν σεβαστοί. Θα πρέπει εμείς να υποστηρίξουμε τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις. Θα πρέπει να κουβεντιάσουμε μαζί με αυτές τις δυνάμεις. Να φροντίσουμε οι φιλοευρωπαϊκές φωνές στη δημοκρατία της Μολδαβίας να ακούγονται. Πρέπει να δράσουμε οι πολιτικές διακηρύξεις δεν αρκούν, χρειάζεται δράση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, σας χαιρετίζω εσάς τους εκπροσώπους των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Συνεχίζοντας τη συζήτηση, δίνω το λόγο στον κύριο Μίξερ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπατικπρόσωπη, η ανατολική γειτονία και η πολιτική όχι μόνο εξυπηρετεί τι χώρε αυτέ, αλλά και την Ένωση. Η πολιτική σταθερότητα και αυξανόμενη ευημερία στι χώρε τη Ανατολική Εταιρική Σχέση μα δίνει ασφαλέστερη και πιο προβλέψιμη γειτονιά και περιορίζει τη δυνατότητα των αντιπαλών μα να ασκήσουν αρνητική επιρροή σε αυτέ τι χώρε. Σαν εισηγητή για τη Γεωργία, συμμερίζουμε τι ανησυχίε για τι εξελίξει σε αυτή τη χώρα. Ε, καταψήφισε το Κοινοβούλιο τη τροπολογία του εκλογικού νόμου που θα είχαν οδηγήσει σε πλήρη αναλογική είναι κάτι ε, που μας λυπεί. Δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε σε εταίρου μας το ακριβές εκλογικό σύστημα που θα πρέπει να χρησιμοποιούν, αλλά προσδοκούμε να συμμορφώνονται από τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι ίδιοι. Οι ευρωπαϊκέ προσδοκίε είναι σχεδόν καθολικά κοινέ για όλους τους πολιτικούς φορείς στη Γεωργία και τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Είναι κρίσιμο να μην αφήσουμε τις θεμητές προσδοκίες αυτές να γίνουν παράπλευρη ζημιά σε, εσωτερικά, σε εσωτερικές πολιτικές Οι ηγέτες στη Γεωργία θα πρέπει να βρουν πολιτική λύση στην κρίση και να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ότι ο λαός τους και οι διεθνείς τους εταίροι θα κινούνται μέσα σε κεραιότητα της πολιτικής διαδικασίας που θα είναι εγγυημένη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, συνάδελφοι, Γκρόσεκ, από το Renew έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η ανατολική εταιρική σχέση είναι στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά το, τους, ε, τις φάσεις εκδρομοκρατισμού, ε, στις περισσότερες χώρες υπάρχουν ολιγάρχες, που είναι κατά των συμφερόντων του λαού και τους απομακρύνουν από τις ευρωπαϊκές αξίες. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται εν κενό και χωρίς την συμμετοχή ξένων παικτών. Η Ρωσία επηρεάζει ανοιχτά και επιθετικά το πολιτικό σύστημα των περισσότερων κρατών στην περιοχή και η Τουρκία δραστηριοποιείται περισσότερο στο να επιδιώκει τα γεωπολιτικά της συμφέροντα και υπάρχει και η Κίνα που ε, δρά πιο κρυφά αλλά και αυτή προκαλεί ζημιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθε η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την ανατολική εταιρική σχέση για να γίνει μεταρρύθμιση και να έχουμε δημοκρατικές ε, δυνάμεις. Ο κύριος ε, Κρασνοδέσκη. Κυρία Πρόεδρε, η ανατολική εταιρική σχέση έχει ε, συνέπειες ε, και έχει αποδώσει γιατί αν κάνουμε σύγκριση με την Μεσόγειο βλέπουμε ότι στέφτηκε από τεράστια επιτυχία αλλά δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στα προβλήματα. Σε κάποιες χώρες της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης έχουμε οπισθοδρόμηση, εκεί εντάσσεται και η γεωργία. Ε, είχαμε την εντύπωση ότι η χώρα ακολουθούσε καλό δρόμο, αλλά αυτά που είδαμε τους τελευταίους μήνες, οι διαμαρτυρίες, η ε, σκληρή στάση της κυβέρνησης, η θέση του κυρίου Γκαχάρικ ο οποίο πριν από λίγο, μέχρι πριν από λίγο ήταν Ρώσο πολίτης και πάρα πολλά άλλα παρεμφερεί. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι στην Αρμενία η πρόοδος οφείλεται στην ανατολική εταιρική σχέση. Ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μας, αλλά η επιτυχία της στρατηγικής εξαρτάται βέβαια και από τη δική μας την αξιοπιστία και από το κατά πόσο είμαστε και εμείς πρόθυμοι να εφαρμόσουμε τα δικά μας τα πρότυπα. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σόκολ έχει μπλε ερώτηση ή απλώς παίζατε με την κάρτα. Τι ακριβώς είναι, θέλετε να κάνετε ερώτηση. Α, ερώτηση θέλετε. Ε, δέχεστε εσείς ε, την μπλε κάρτα από τον κύριο Σόκο. Κύριε Κρασοντέψκη. Would you accept a blue card from... Da? Δέχεστε μπλε κάρτα. Ε, δέχεστε. Οι χώρες αυτές, μερικές εξ αυτών, έκαναν βήμα προς τα πίσω όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε αρκετά για να τις βοηθήσει. Ήταν αρκετά συνεπής στο να στηρίξει τις χώρες αυτές. Και πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ενιαία πολιτική και μπορεί να στηρίξει αυτές τις χώρες. Για ένα λεπτό η απάντηση. Ε, γι' αυτόν ακριβώ